Ε, good afternoon, um, everybody. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, λέει η Πρόεδρος. Καθίστε να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Έχουμε την τιμή να αρχίσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση για ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Μοσκοβισή. Δεν έχουμε θεία αρκετό καιρό, αλλά χαιρόμαστε που τώρα ήρθατε Οπότε θα ήθελα να επενθυμίσω ότι σήμερα θα συζητήσουμε για την ε, πρόοδο στο πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το σχέδιο διαχείρισης 17 για την πολιτική που αφορά τα τελωνία, αλλά θα συζητήσουμε και τις μελλοντικές πρωτοβουλίες. Ε, επίσης, να συζητήσουμε για την ε, πρώτα του νομοθετικού έργου, ότι ήδη έχει παρουσιάσει η Επιτροπή, αλλά για κείμενα που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί. Ίσως ε, επίσης να ανταλλάξουμε απόψεις όσον αφορά τις προτεραιότητες για την περίοδο 2017-2018. Με αυτή την σύντομη εισαγωγή ήρθε η ώρα να σας δώσουμε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Αντιπρόεδρε, βουλευτές. Πρώτα-πρώτα συγχαρητήρια για την εκλογή της Προέδρου. Όντω δεν τα έχουμε βγει εδώ και ε, πολύ καιρό, αλλά είχα άλλε ε, ποικίλε υποχρεώσει. Ε, έχουμε και την πρωτοβουλία για την Τελωνιακή Ένωση. Πρώτα-πρώτα, ξέρετε το, το πόσο έχουν τεχνικό χαρακτήρα και τεχνοκρατικό τα θέματά μας, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά σε πολλά επίπεδα. Και πρώτα-πρώτα και σας τονίζω ότι πάντοτε προβάλλονται ότι αυτό είναι σημαντικό εργαλείο κατά της τρομοκρατίας, κατά της, χρηματοδότηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όσον αφορά τον έλεγχο ε, υγειονομικών και διατροφικών ειδών. Όλα αυτά γίνονται από τα τελωνία και δεν αξιολογείται πάντοτε και δεν εκτιμάται αυτό. Και επίσης ε, έχουμε τη διερεύνηση των, ε, εμπορικής μας και της εμπορικής μας οπότε επίσης έχουμε και την αξιακή παγκόσμια αλυσίδα που έχει οικονομική σημασία και οπότε χρειάζεται ένα τελωνιακό σύστημα αποτελεσματικό. Και πρόσφατα όλα αυτά προβλήθηκαν σε αυτή μας τη συμφωνία, την στρατηγική με την Κίνα. Πριν από λίγε εβδομάδες μόλις, επί τη ευκαιρία της συνάντηση κορυφής με τη χώρα εκείνη. Και ε, επίσης, μέσω του εμπορίου ε, προβάλλουμε τι αξίες μας κόντρα στους φραγμούς και στον προστατευτισμό οπότε και αυτή μας η τελωνική δράση αναδεικνύει την προτεραιότητά μας για το να υπάρχει ένας άλλος δρόμος, δρόμος των ελευθέρων συναλλαγών υπό έλεγχο. Ε, επίσης, τα, η τελωνική πολιτική είναι στοιχείο ανταγωνιστικότητας. Και με μια μελέτη μας είδαμε ότι η τελωνία ήταν ένας από τους χειρότερους εφιάλτες, τους 10 τους εφιάλτες των ΜΜΕ και οι επιχείρησει που μπορούν να χειριστούν τελικά θέματα και κερδίζουν χρόνο, άρα μεγάλη σημασία. Είναι επομένω ε, το τελωνίο ένας ε, καταλήτη εξυγχρονισμού τη δημοσιακή πολιτική για απλούστευση, για την αποϊλοποίηση των συναλλαγών, για την ε, αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών, αυτοματοποίηση κλπ. Είναι μια ήσυχη επανάσταση που γίνεται εδώ και χρόνια στα τελωνία. Και ε, τα έχουμε δει αυτά. Από τότε που ανέλαβα τα καθηκοντά μου στην Γαλλία. Και είδαμε ότι πρόκειται για ένα εργαστήρι εξυγχρονισμού όσον αφορά την ε, κρατική διοίκηση. Και για τα κρατημέλη, για εσά και για μας υπάρχει και η δημοσιονομική διάσταση είναι η οικονομική πόρη που είναι αρκετά σημαντική. Σήμερα και όλα στο πρωί τα συζητήσαμε για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε βοηθούν τα τελωνία για τις σχέσεις μας με τον εξωτερικό κόσμο. Έχουμε τις σχέσεις με την ε, Τουρκία που είναι στο επίκεντρο της προσοχής. Έχουμε συνεχή συνεργασία με τη χώρα εκείνη ε, πρέπει να επαναορίσουμε τη σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και η τελειωνιακή διάσταση επομένως έχει στρατηγική σημασία και για το Brexit. Να, ποιο είναι το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο της ε, πρωτοβουλίας μας. Επομένως δεν είναι μόνο τεχνική διάσταση του θέματος, αλλά είναι πάρα πολύ πολιτική. Οπότε για την σχετική διακυβέρνηση βλέπετε ότι έχουν πρωτοβουλίε που ανταποκρίνονται στη δύο σα ψηφίσματα. Ε, αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν ω αφετηρία το ότι θέλουμε να ενεργούμε, να δρούμε ε, σε βάση συνεργασίας για όλα τα επίπεδα μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεργασία. Να υπάρχει αυτή η στρατηγική οπτική, ε, αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας, ε, συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ούτως ώστε να υπάρχει μια υποστήριξη λειτουργική, επιχειρησιακή, συνεργασία μεταξύ τελωνίων και άλλων αρχών, ούτως ώστε να υπάρχει ανάκτηση των ε, πόρων, επίσης συνεργασία με τους ε, οικονομικούς παράγοντες, γιατί και εκεί υπάρχουν κάποιες προκαταλήψεις και όλα αυτά να κατατείνουν σε καταλήτη κομπής δραστηριότητα. Και έχουμε δεσμευτεί προς Συμβούλιο και Κοινοβούλιο να κάνουμε μια έκθεση ανά διετία και αυτή η έκθεση θα έχει δύο στόχους. Πρώτα-πρώτα θα ενημερώνει, θα συμπληρώνει τα σχετικά με την εφαρμογή του τελωνιακού κώδικα, όπως έλεγε και το δικό σας ψήφισμα. Στρατηγική μαζί με τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες. Δεύτερος στόχος είναι το να έχουμε κάποιο είδους δίκτυ, κριτήριο της ε, απόδοσης και επιδόσεων της κοινωνική πολιτικής. γιατί αυτό είναι το πρώτο το οποίο δουλεύουμε. Δηλαδή να υπάρχει αυτό το, αυτή, αυτή η σειρά των κριτηρίων, ούτω ώστε να ξέρουμε πώ θα λαμβάνουμε αποφάσει και πώ θα χαράσουμε μια στρατηγική και ένα σχέδιο δράση, λαμβάνοντα υπόψη του κινδύνου, αυτά τα οποία έχουμε ήδη πει για την αποτελεσματικότητα τη πολιτική μα και επίση, κατά τρίτον, θέλουμε να εξασφαλίζουμε την ενιαία ερμηνεία του τουλιανικού δικαίου, την ομοιόμορφη ερμηνεία σε όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε ακόμη υπάρχει ε, πανσπερμία ερμηνεών του Τελωνικού Κώδικα. Ε, δεν έχουμε πάντα τους ίδιους ε, κανόνες του παιχνιδιού. Αυτό είναι παράδειγμα γιατί θεμέλιο της Ένωσης είναι η ιστορική αγορά. Οπότε πρόκειται εμείς να εκπονήσουμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας σε συνεννόηση με τα κράτη-μέλη και τους οικονομικούς παράγοντες. Και όπως είπαμε αυτοί ε, σας απασχολούν πολύ συχνά και οπότε θα συμμετάσχουν πλήρως στο έργο, στην προσπάθειά μας και εμείς δεσμευόμαστε να αναβαθμίσουμε τους υπάρχοντες μηχανισμούς της διαβούλευσης με αυτούς. Έχουμε και την ομάδα επαφής με αυτούς τους οικονομικούς ε, παράγοντες και σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις και τη διοίκηση. Επίσης θα κοιτάξουμε και για το σύστημα πληροφορικής, το οποίο επίσης σας ενδιαφέρει. Είναι κλειδί αυτό, ούτως ώστε να διχίσουμε τους κινδύνους, άρα και την ασφάλειά μας. Οπότε θα πρέπει να γίνει ε, προβληματική σε, σε βάθος και έτσι να έχουμε ένα τέτοιο πολιτές πλαίσιο. Δεν αντιλαμβάνονται όλα τα κράτη με τον ίδιο τρόπο το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το κοινό σύστημα πληροφοριών. Αλλά αυτό εξυπηρετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να συνδέεται με τα εθνικά συστήματα μέσα στα πλαίσια των δημοσιογών περιορισμών που γνωρίζουμε. Επομένω, είναι δυτή η προσπάθειά μα. Πρώτα-πρώτα, μακρόπνο σχέδιο για τι ε, υποδομέ πληροφορική, να δούμε ε, το πώ θα έχουμε προσθέμενη αξία και επίση θέλουμε να υπάρχει συνέργεια με τις ε, υπάρχουσες υπηρεσίες διαχείρισης ε, πληροφορικής και πληροφοριών. Επίσης, θέλουμε να αναβαθμιστεί η συνέργεια με τις υπόλοιπες διοικήσεις και κυβερνήσεις. Επίσης, ε, κατά της εγκληματικότητας, συνεννόηση με τις αρχές όσον αφορά την διαχείριση των συνόρων, ακριβώς, και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής συνεργαζόμαστε και με τις φορολογικές αρχές ε, όσον αφορά την ίσπραξη του ΦΠΑ και τα σχετικά με τα εμπορεύματα και βέβαια η πόρη από τον ΦΠΑ είναι μια βάση, ένα θεμέλιο για τους ιδίους πόρους στην Ευρώπη και αυτό επίσης είναι μεταβλητή σημαντική και παράγοντα που λαμβάνει την υπόψη για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και βέβαια κύριε Πρόεδρε θα συνεχιστεί και με τη δική σας Προεδρία η αγαστή συνεργασία μας. Όπως και εσείς και εγώ πιστεύω ότι το τελωνίο είναι υπόθεση πολύ σημαντική για την Ευρώπη και απαιτείται συνεργασία και απαιτείται και πίεση με την καλή έννοια από πλευράς μας για να κάνουν τα προόδου τα κρατημέλη, αλλά και η Επιτροπή. Άρα χρειάζεται αυτού του είδους η διαλεκτική σχέση μεταξύ μας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, θα... Είναι δύσκολο να αλλάζει κανείς γλωστές. θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στους συντονιστές των διαφόρων πολιτικών ομάδων αν θέλουν να, έχουν, αν θέσουν κάποιο ερώτημα προς τον Επίτροπο, ο Ανδρέας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Χαίρομαστε ιδιαίτερως ε, που βρήκατε το χρόνο σήμερα να ήλθετε στην Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα ζητήματα τα οποία θέσαμε στην Ολομέλεια και τα οποία απασχολούν πολλούς ε, συναδέλφους ε, μας ανησυχούν και μας κάνουν άκρος επικριτικούς και νευρικούς. Γιατί, διότι έχουμε την εντύπωση ότι ο Ευρωπαϊκός Τελωνιακό Κώδικας ε, κινδυνεύει να μην εφαρμοστεί όπως εμείς θα θέλαμε. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις ε, και νομίζω ότι στην εισαγωγική σας παρέμβαση ακροθικώς αναφερθήκατε σε αυτά τα θέματα, θέλω όμως να εμβαθύνετε λίγο παραπάνω. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι σε αυτό το πλαίσιο νομίζω πρέπει να ξαναπούμε ότι ξεκινήσαμε μια διαδικασία ε, ήδη από το 2005 για να νομοθετήσουμε για τα θέματα αυτά, πολύ πρέπει να αναλάβετε εσείς το χαρτοφυλάκιο αυτό. Αποτύχαμε νομίζω το 2011 με τον εξεχρονισμένο τελωνιακό κώδικα νέα απόπειρα. Τώρα ελπίζουμε αυτή να λειτουργήσει. Όπως είπατε όμως, στα ψηφιακά συστήματα που θα πρέπει να δημιουργήσουν τα κράτη-μέλη, ακόμα είμαστε σχεδόν στο τίποτα. Ε, δεν έχουν κάνει σχεδόν τίποτα ακόμη δηλαδή τα κράτη-μέλη. Και είναι προφανές ότι 7 στα 28, σε ό,τι αφορά το 100% των τελωνιακών εξόδων, το κατάλληλο δεν έχουν ακολουθήσει αυτό που προτείνετε εσείς πέραν των οικονομικών πόρων. Τι προτείνετε σε σχέση με την υποδομή πληροφορικής για τον τελωνιακό κώδικα. Να μην καθυστερήσει κι άλλο. Μήπως με κάποια οικονομική υποστήριξη ε, με ευρωπαϊκά κονδύλια θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη. Και δεύτερον, από νομική πλευρά τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακόμη για να τα ξεπεράσουν. Θα γνωρίζετε ίσως ότι στη δική μας Επιτροπή μπορούμε να ακολουθήσουμε την ταχεία διαδικασία μόνο εάν δεν υπάρχει ούτε ένα κράτος μέλος που να εναντιωθεί σε αυτήν. Έστω και έναν εναντιωθεί δεν μπορούμε να την ακολουθήσουμε. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Concerned... Ανησυχώ. Ανησυχώ ότι δεν θα τεθεί σε εφαρμογή ο τελωνιακός κώδικας εγκαίρως. Και θα είναι η δεύτερη αποτυχία μας. Ευχαριστώ. Εσείς έχετε ερωτήσεις. Νίκολα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Επίτροπε. Καλώς ορίσατε. Είναι σημαντική αυτή η συνάντησή μας. Θα ήθελα να, να δούμε κάποια άλλα πράγματα, έτσι, δευτερεύοντα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα θέματα τα τελεμιακά. Είναι στρατηγική σημασία για την ε, μέρημνα μα, για την εσωτερική αγορά, για την εύρυθμη λειτουργία τη όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο. Είναι στρατηγική σημασία, ακριβώ όπω ε, το αναδείξατε στην ομιλία σα. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Πρώτα-πρώτα, έχουμε την ε, οδηγία εκείνη που αφορά τις κυρώσεις όσον αφορά τις ελληνικές παραβάσεις του Συμβουλίου. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ε, ληφθεί κάποια μερίμνου ώστε να αρθεί αυτό. Είναι ένας φραγμός. Η Όλαφ, όπως λέει και ο Διεθνής Τύπος, πριν από λίγες εβδομάδες, πριν από λίγους μήνες ανακάλυψε μία απόλαψη, αποφυγή καταβολής κάποιων δασμών αξίας δισεκατομμυρίων. Και αυτά αφορούν τον, τομέα, τον κατασκευαστικό, ε, στον τομέα των κλωσφαντουργικών στην Ευρώπη. Ε, αυτά είναι θέματα τα οποία, στα οποία έχουμε ευαισθησία, αλλά θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Και εμείς προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί κατεπηγόντως πρέπει να τα διαχειριστούμε αυτά. Συμφωνούμε πάρα πολύ με αυτά που είπατε και ακριβώ όπω είπατε ότι δεν θα πρέπει να υψώνουμε ε, τείχους, ε, ακριβώ όπω κάνει όπω είπατε και η Αμερική τα τείχη του Ατλαντικού. Αυτό πάνε να πει εμπόριο για μα. Ε, οπότε κύριε Επίτροπε, σήμερα χρειαζόμαστε επίγουσε απαντήσει για το θέμα αυτό. Πώ δηλαδή εμεί μπορούμε έστω και σε στενά χρονικά πλαίσια να ε, ε, θεσπίσουμε κάποιους ε, κανόνε ούτω ώστε να καταπολεμήσουμε την παραποίηση, τι απομιμήσει που χτυπάει την οικονομία μα και έχει στριμώξει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you very much, Nicola. And then e και για το ECR. Ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε κύριε Επιτροπέ. Θα ήθελα ε, να συζητήσουμε κάποια ε, ναι. θέματα αφενός. Ε, τα τις αποστολές χαμηλής αξίας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει η εκτελεστική, η πράξη ε, που παραμένουν σε μια μεταβατική περίοδο, όμως τα ταχυδρομεία έχουν αυτό το ε, δικαίωμα και έχουμε αυτή την ασυμμετρία λοιπόν. Γνωρίζω ότι η Κομισιόν προσπαθεί να ξεκινήσει ένα, ε, ένα καινούριο πρόγραμμα. Το ερώτημα μου είναι πώς προχωρά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, διότι από την πλευρά των καταναλωτών πολλές φορές οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τι διαφορέ και τα κόστη που προκύπτουν από αυτά. Το δεύτερο θέμα το οποίο θα ήθελα να, να συζητήσουμε αφορά τις αποστολέ χαμηλή αξία όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ε, υπάρχουν πολλοί ψηφοφόροι μου που επικοινωνούν μαζί μου και ε, ε παραγγέλνουν πράγματα από εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα από τι ιστοσελίδε των ΗΠΑ κάτι το οποίο κοστίζει 150 ευρώ για παράδειγμα, τότε ε, ε, στα τελωνία σταματάνε την εισαγωγή, ε, παίρνουν ένα πρόστιμα, ε, λαμβάνουν ένα, ε, μία επιστολή από τις τελωνιακές αρχές οι οποίες δεν μπορούν να κάνουν τη διαφοροποίηση Οπότε ε, σε αντιμετωπίζουν ε, σαν επιχείρηση, πρέπει να πληρώσεις ε, φόρο, πρέπει να τιμωρείς, οπότε υπάρχει και το κοιτάω αυτό στο πλαίσιο του Brexit, διότι αυτή τη στιγμή είμαστε στην Τελωνιακή Ένωση και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να παραμείνουμε. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι σε περίπτωση που δεν είμαστε, τότε υπάρχουν πάρα πολλές, ε, ε υπάρχει εμπόριο μεταξύ μας, ε, ε, δώρα για παράδειγμα, ε, και θα ήθελα να ρωτήσω αν η Κομισιόν έχει σκεφτεί στο ζήτημα της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και γενικότερα όσον αφορά το διεθνές εμπόριο τι θα γίνει με αυτούς τους κανονισμούς διότι ιδάλλως ε, το ηλεκτρονικό εμπόριο το, για, τους, για τους μας είτε σε εισαγωγές είτε σε εξαγωγές επηρεάζεται από αυτός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. και η ΚΑΙ από την άλλη. Ευχαριστώ. Έχουν ε, γίνει ε, πολλές συζητήσεις σχετικά με την Τελωνιακή Ένωση ε, και για να έχουμε μια ε, τελωνιακή ένωση που λειτουργεί. Το σημαντικό είναι ε, να έχουμε και ένα πανευρωπαϊκό ηλεκτρονικό τελωνιακό σύστημα όμως από ό,τι ακούω υπάρχει μια καθυστέρηση στην εξέλιξη αυτού και αυτό ίσως να καθυστερήσει την εφαρμογή του ενωσιακού τελωνιακού κώδικα. Το ερώτημά μου είναι ποιες συγκεκριμένες δράσεις σκοπεύει να αναλάβει η Κομισιόν νησιών ώστε να έχουμε ε, ένα ενοποιημένο ε, σύστημα ε, πληροφοριών και δεύτερον τι θα κάνει η Κομισιόν για να μπορέσει να διασφαλιστεί ότι θα εφαρμοστεί εγκαίρως ο ενωσιακός τελωνιακός κώδικας και το άλλο θέμα αφορά τις κυρώσεις και τις διαδικασίες επιπαραβάση τις οποίες ανέφερε ήδη ο συνάδελφος κύριος Ντάντε κάναμε την έκθεση εδώ ε, και θέσαμε την ε, θέση του Κοινοβουλίου. Γνωρίζουμε ότι η πρόταση αυτή έχει κολλήσει στο Συμβούλιο. Κατανοώ λοιπόν ότι η Κομισιόν δεν αποσύρει την πρόταση, όμως ε, ποια είναι τα επόμενα βήματα, ποια είναι η ιδέα, πώς θα προχωρήσουμε με αυτό, τόσο ώστε να έχουμε ένα ενοποιημένο σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και ο Ντένις μου από την ΚΟΥΕ Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, επειδή δεν ήμουν το πρωί εδώ, ε, συγχαρητήρια με την εκλογή σου ως ε, πρόεδρος της Επιτροπής μας. Έχω τρία σημεία. Το ε, πρώτο αναφέρθηκε από την πλευρά της Άλντε. Θεωρώ ότι όλος ο εξυγχρονισμός του ενωσιακού τελωνιακού κώδικα στόχευε το να έχουμε ένα κεντροποιημένο σύστημα, ένα τεχνολογικό σύστημα το οποίο θα λειτουργεί. Ε, και ε, μαθαίνω και εγώ όπως οι άλλοι ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, ότι διαρκεί πάρα πολύ και όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να αποτύχει επειδή δεν έχουμε την τεχνολογία για όλο αυτό. Ε, έτσι λοιπόν, Επίτροπε, σας παρακαλούμε επιταχύντε το. Το δεύτερο θέμα αφορά την, τον εγκεκριμένο οικονομικό φορέα. Υπάρχουν πάρα πολλές διαδικασίες ε, για να ε, γίνει κάποιος συγκεκριμένος οικονομικός φορέας, ε, για να, έχει, για να έχουμε λιγότερους ελέγχος για τα αγαθά τα οποία εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως ε, αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι ε, βασίζεται στις συναλλαγές και όχι στην επεξεργασία ε, με αποτέλεσμα η προστιθέμενη, η προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο θα ενισχύσει την κατάσταση για τους εγκεκριμένου οικονομικούς φορείς, ε, για τις απλοποιημένες διαδικασίες, όμως ταυτόχρονα βλέπουμε και θα πρέπει να ομολογήσω ότι και στη χώρα μου υπάρχουν περιπτώσεις ε, διαφθοράς της τελωνιακής υπηρεσίας, οπότε χρειάζονται και κάποιοι έλεγχοι στην κυβέρνηση για να ε, διασφαλιστεί η φερικαιότητα. Το ερώτημα ε, μου λοιπόν είναι αν το πιλωτικό πρόγραμμα θα αρχίσει ε, και θα ε, συγκεράσει αυτό το δύο περισσότερες πολιτικές για την φερεγγιότητα και πιο απλές διαδικασίες για τους συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς και σε περίπτωση που το πολιτικό πρόγραμμα λάβει η χώρα στη συνέχεια θα ήθελα να ρωτήσω αν η Κομισιόν μπορεί να συμμετάσχει και να κάνει ελέγχους είναι απλά ένα ε, project στο τέλος ε, του οποίου θα ε, δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Και το τελευταίο σχόλιο είναι ότι ακούω από την, οικονομική, από την επιχειρησιακή κοινότητα είναι ότι το έργο της Κομισιόν είναι καλό, περισσότερο από, καλύτερο από ό,τι περιμένουμε από αυτή την Επιτροπή. Ε, για νομική βεβαιότητα λοιπόν θα μπορούσατε να δώσετε αυτές τις κατευθυντήριε, οι οποίες θα είναι νομικά δεσμευτικές ούτω ώστε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τα ίδια πρότυπα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον Τενίστε Γιόγκ, η Άννα Μαρία. Σε ευχαριστώ, Ανελίν. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο, τον οποίο θέλω και να καλωσορίσω. Αυτά που είπατε για την σιωπηρή επανάσταση, την τελωνιακή και για τη σημασία του τελωνιακού τομέα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ε, είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπατε για το Brexit, ε, τη μεταρρύθμιση. Για την Τουρκία και τη Συμφωνία Εταιρική σχέση. θα ήθελα να μου πείτε και πώς θα καταπολεμήσετε την απάτη και τις παρατυπίες και θα έλεγα επίσης εγώ και τα παραποιημένα τα τρόφιμα, τις απομνήσεις. Θα, θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας σε σχέση με τα ψηφιακά βιβλία. Τι έγινε στο Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς ε, είχαμε ψηφίσει 590 υπέρ το Μάιο τη δυνατότητα εναρμόνισης δηλαδή να είναι το ίδιο το καθεστώς ΦΠΑ για τα ηλεκτρονικά ψηφιακά βιβλία, αλλά το θέμα έχει κολλήσει στο Συμβούλιο. Με αποτέλεσμα να έχουμε τον το συντελεστή ΦΠΑ 15% και 5% είναι για τα έντυπα. Πού είναι η ψηφιακή επανάσταση και πώς θέλετε να προχωρήσουμε πάνω στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ την Αννα Μαρία. Η Μαρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Μπορώ να μιλήσω και τη γλώσσα μου. Α, τέλεια. Μεταφράζεται. Μεταφράζεται, μεταφράζεται. Υπήρξε μια προσπάθεια να εφαρμοστεί αυτό το σύστημα στα κράτη-μέλη και το 2016 αλλά υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση σε πολλά κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τελικά το κατά πόσον ε, τα συστήματα πληροφορικής ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφαρμός, εφα, ε, επαρκώς. Υπάρχει και το θέμα της μείωσης του κόστους. Θέλουμε όμως να μειωθούν και κίνδυνοι για την κοινωνία. Το 2007, 30 Μαΐου, η ομάδα ηλεκτρονικού συντονισμού ε, έχει δημοσιεύσει κάποιες μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες θα ισχύουν το 2020. Δεν ισχύουν όμως ήδη πλέον. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε ως πρόθεσμα το 2020 πια και τι πρέπει να γίνει αν θέλουμε να υπάρχει ασφάλεια και επιχειρηματική ασφάλεια και ασφάλεια τους πολίτες. Σίγουρα θέλουμε να διευκολύνουμε το εμπόριο, αλλά τι θα γίνει μέχρι το 2020. Μην έχουμε ακόμη καθυστέρηση 3, 4, 5 χρόνια. Αυτά θα ήθελα να σας ρωτήσω. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Εύαν Στέφανεκ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τι που μας έδωσε. Είπατε ότι υπάρχει ανάγκη για ίδιου πόρους και συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Στηρίζω το στόχο της Κομισιόν για τους ίδιους πόρους. Ταυτόχρονα όμως γνωρίζουμε ότι η φορολογία είναι εθνική αρμοδιότητα. Και υπάρχει η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί να μην αυξηθεί το φορολογικό άρθρος για επιχειρήσεις και φορολογουμένου. Πώς μπορείτε λοιπόν να φροντίσετε εσείς να έχουμε μεν ιδίους πόρους, αλλά να μην αυξηθεί η φορολογία συνολικά από την άλλη. Ευχαριστώ λοιπόν πρόεδρο. Κάποιος άλλο θα ήθελε το λόγο, ενδεχομένω, να θες κάποιο ερώτημα, αν όχι τότε... Θα ήθελα και εγώ, αν μου επιτρέπετε, να σα κάνω μια ερώτηση η οποία έχει να κάνει με αυτό που είπε η κυρία Γκραπίνη για τα συστήματα πληροφορικής που δεν είναι επαρκή και πώς θα εγκαιθούμε την ασφάλεια των πολιτών αφού δεν είναι επαρκή και δεύτερον σε ό,τι αφορά τον Brexit έχω ένα ερώτημα. Ελπίζουμε φυσικά να υπάρξει ένα είδος τελωνιακής ένωσης ή κάτι τέλος πάντων ε, με, το Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως η Ευρωπαϊκή Τελωνιακή Ένωση πώς θα αντιμετωπίσει τη μεγάλη ροή ε, προϊόντων από το Ηνωμένο Βασίλειο και Τούμπαλιν. Παρακαλώ να απαντήσετε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να δώσω στο δυνατό περισσότερες απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα, πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εφαρμόσει το σύστημα πληροφορικής. Και τι θα συμβεί αν υπάρξουν καθυστερήσεις. Γνωρίζουμε ότι μέχρι το 2020 πρέπει να έχουν εφαρμοστεί όλα αυτά τα συστήματα πληροφορική για τον ελληνικό κόσμο. Κατόπατε αρκετοί από εσά και σίγουρα οι πιέσει ε, στα κράτη-μέλη είναι μεγάλε, αλλά και στην Κομισιόν και στο εμπόριο που οι κλάδοι διάφοροι μα έχουν ενημερώσει ήδη για τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αναλύει πολύ προσεκτικά από κοινού με τα κράτη-μέλη το κατά πόσο είναι εφικτό να λειτουργήσουν αυτά τα συστήματα και ποιε θα είναι οι νομικέ συνέπειε σε περίπτωση καθυστέρηση. Παρότι θεωρούμε ότι τα περισσότερα συστήματα πληροφορική θα είναι έτοιμα το 2020 και θα είναι ε, λειτουργικά. Αυτή είναι η προθεσμία καταληκτική, όπω ξέρετε, το 2020 δηλαδή. Ένα άλλο ερώτημα, αν κατάλαβα καλά, ήταν να σας περιγράψω την πρόοδο και ο κύριος Φαπ νομίζω το έθεσε. Σε σχέση με την αρχιτεκτονική, την εθνική, θα πρέπει σιγά σιγά να αντικατασταθεί. Η δουλειά για τα συστήματα αυτά της πληροφορικής ξεκίνησε το 1998 με τα νέα μηχανοργανωμένα συστήματα διαμετακόμισης, το CPS που εγκρίθηκε το Έκτοτε αναπτύχθηκαν πολλά άλλα συστήματα και μέχρι τώρα λειτουργούν καλά. Τα 17 συστήματα πληροφορικής έχουν αναβαθμιστεί πολλές φορές και έχουμε και νέα φιλόδοξα project όπως ατελωνικές αποφάσεις με ευρωπαϊκή ισχύ, διασάφηση κεντρωτική, κεντρική κτλ. κτλ καταληκτική προθεσμία για την ολοκλήρωση των συστημάτων πληροφορική είναι το 2020. Πάντοτε ξέραμε ότι τα φιλόδοξη η προθεσμία λόγω των πολύ σημαντικών αλλαγών και του τεράστιου φάσματος που πρέπει να καλυφθεί. για την ανάπτυξη των διαφόρων συστημάτων. Και η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα η εναρμόνιση για τη διελειτουργικότητα και ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις για την αναβάθμιση των συστημάτων. Σε ό,τι αφορά τον αυτοματισμό του τελεινικού περιβάλλοντος, την μηχανοργάνωση δηλαδή, έχουν γίνει πολλά είδη. Περί αναβαθμίσεων ουσιαστικά πρόκειται, είτε υφιστάμενων συστημάτων, είτε συμπλήρωση ε, των υφιστάμενων εφαρμογών. Βέβαια, απομένει ακόμη να γίνει κάποιο έργο. Πρόοδος πάντως έχει σημειωθεί, τα αναλύουμε όλα αυτά και θα σας ενημερώσουμε εκ νέου για τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών. Πώς σκοπεύει η Κομισιόν να αντιμετωπίσει την απάτη ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τα τελωνιακά. Ήταν μια ερώτηση. Έχουμε την διαδικασία 42, όπως λέγεται, Procedure 42. Ξέρουμε τι κάνουν ορισμένα εγκληματικά δίκτυα που εισάγουν ε, προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί να πληρώνουν στην χώρα πώληση ε, τον ΦΠΑ. Αυτέ οι ομάδε ουσιαστικά κερδοσκοπούν ε, στι πλάτε των Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα σα επαναλάβω, ότι επί σειρά ετών τώρα τονίζει ότι θα πρέπει να ελέγχονται καλύτερα εισαγωγές και θα πρέπει να βλέπουμε πού ε, πηγαίνει η πρόσοδη αυτών των ε, συναλλαγών γιατί καλύτερα να εντοπίσουμε ταχύστα την απάτη του ΦΠΑ, ώστε να μην μπορούν οι ομάδες αυτές να συνεχίζουν ανενόχλητες και χωρίς επιπτώσει τη δράση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Φορολογικές διοικήσεις ε, θα πρέπει και τελωνιακές αρχές να συνεργάζονται. Και αυτό θα πλουστεύσει και τη ζωή των επιχειρήσεών μας στην νέα αγορά. Αυτό που επίσης θέλουμε να διευκολύνουμε, το είπε και ο κύριος ε, Ντάντι, είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο, το e-commerce, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Η Κομισιόν λοιπόν θεωρεί ότι θα πρέπει να διευκολυνθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ταυτόχρονα Είχαμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις, τα παραποιημένα προϊόντα, μιμήσεις. Όλα αυτά πολλαπλασιάζονται. Πρέπει λοιπόν μεν να διευκολύνουμε το εμπόριο, αλλά να προστατεύσουμε και τα έσοδα. Καθώς επίσης και την ασφάλεια, την ακαιρεότητα, τα δικαιώματα και το ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ εμπόρων από Ένωση και εκτός Ένωσης συνεργαζόμαστε, υπάρχουν πλατφόρμες, υπάρχουν διάμεσοι φορείς και διεθνείς οργανώσεις με τους οποίους έχουμε επαφές για να μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή εποπτεία του εμπορίου χωρίς να παρακολύουμε τη ροή αγαθών. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Είχαμε πρόσφατα την πρόταση για το ΦΠΑ και αυτό μαζί με την πλήρη εφαρμογή του τελωνιακού κώδικα θα παράσχει μία μακροχρόνια λύση για τις αλλαγές αυτές που μπορεί να φαίνονται ουσιαστικά αντιφατικές μεταξύ τους. Η Όλαφ έκανε μία έρευνα για τις αγωγές αγαθών ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε σχέση με τη διαδικασία 42, κατά πόσο υπάρχει απάτη ΦΠΑ κτλ. Η τελευταία σχετική έρευνα της Όλαφ δείχνει ότι συνεχίζεται εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια το φαινόμενο αυτό, χωρίς να υπάρχουν συνέπειες. Αν αυτοί οι ισχυρισμοί, αν οι καταγγελίες αυτές επιβεβαιωθούν, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα αγαθά ουσιαστικά ε, πηγαίνουν ε, στην παραοικονομία. Αυτήν την ε, οικονομία, την παραοικονομία τροφοδοτούν. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την απάτη με το ΦΠΑ και είναι μεγάλη προτεραιότητα για την Κομισιόν. Ξέρετε ότι το φθινόπωρο θα σα παρουσιάσω μια φιλόδοξη πρόταση για την μεταρρύθμιση του παροχημένου καθεστώτο ΦΠΑ. Και εδώ να απαντήσω και στην κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Επειδή σχετίζεται. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και ε, κάποιους κατέβασε μια λογική πρόταση κατά την άποψή μου. Δηλαδή τα κράτη-μέλη να είναι ελεύθερα να ορίζουν μειωμένου συντελεστέ ΦΠΑ για ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις και e-book, e-books, ε, ηλεκτρονικά βιβλία. Εγώ μπορεί να προτιμάω τις ε, έντυπες εφημερίδες και τα βιβλία σε χαρτί, αλλά η εφημερίδα στο διδίκτυο είναι με εφημερίδα. Και το ψηφιακό ηλεκτρονικό βιβλίο είναι βιβλίο, όπως και αν το κάνουμε. Άρα θέλαμε να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ των δύο μορφών. Ουσιαστικά παντού αυτό είναι αναγνωρισμένο από όλα τα μέλη του Συμβουλίου και αυτές οι προτάσεις ε, ε, φαίνεται ότι είχαν οριμάσει για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Τι έγινε όμως, ο νέος Τσέχος υπουργό αρνήθηκε. Και πρέπει να πω εδώ ότι ουσιαστικά ε, ήταν εντελώς ανενημέρωτος, δεν είχε ιδέα του, του θέματος. Κάτι έλεγε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, ε, μια παρέκκληση για το διασυνορικό ΦΠΑ ή Κομισιόν. Δεν είναι αντίθετη, για να σα πω κιόλα την αλήθεια, σε μια τέτοια παρέκκληση, χωρί να θέλουμε βέβαια αυτό να γίνει μόνιμο καθεστώ ή κοινό καθεστώ. Γιατί δεν είναι αυτό ο σωστό τρόπο για να αντιμετωπιστεί ο διασυνοριακό ΦΠΑ και να αντιμετωπιστεί η απάτη με αποτελεσματικό τρόπο στην εσωτερική αγορά. Τώρα, από τον Ολλανδό Υπουργό, τον συνάδελφό μου, τον εξαίρετο συνάδελφο Γερούν Ντάισελμπλουμ, ε, πυροδότησε μία έντονη αντίδραση. Και το καταλαβαίνω. Μιλάμε για μία οικονομία που χαρακτηρίζεται από την ελευθερία. Στην επικοινωνία, στην ενημέρωση. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε δικαίωμα όταν υπάρχει τόσο μεγάλη συμφωνία να μπλοκάρουμε μια τέτοια απόφαση. Γι' αυτό λοιπόν μπορώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν προτίθεται να επιτρέψει να αναβαγίσει η προσπάθεια αυτή. Και μάλιστα ερχόμενος εδώ δέχτηκα κλήσεις από εφημερίδες που μου λένε ότι η οικονομία των έντυπων μέσων ενημέρωση εξαρτάται, η επιβίωσή της εξαρτάται από αυτό το μέτρο. Αν όμως η στρατηγική μας είναι, επειδή έχουμε κάπου αλλού πρόβλημα, να μπλοκάρουμε ένα άλλο ε, θέμα, τι να πω. Δεν με βρίσκει σύμφωνο ούτε με αυτήν την ιδιότητα, ούτε με τις άλλες ιδιότητες που είχα. Είτε στην Επιτροπή, είτε εδώ, είτε στο Εθνική ε, Βουλή δεν θα περάσει. Έτσι. Και έρχομαι τώρα. Συγγνώμη, αυτό έχει να κάνει το πρώτο θέμα. Λοιπόν, έρχομαι πάλι στο πώς μπορούμε να έχουμε διαλειτουργικά συστήματα πληροφορικής. Εμείς εργαζόμαστε με τα κρατη για την εξορθολογισμό, την ευθυγράμμιση της πλήρους, μηχανοργάνωση. πλήρους μηχανοργάνωσης των διαδικασιών ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τα συστήματα πληροφορική για τα τελωνία στο εθνικό περιβάλλον πληροφορική με κοινό τρόπο. Έχουμε ένα κοινό μοντέλο δεδομένων, το οποίο φεγγραμμίζεται με το διεθνές μοντέλο του παγκόσμιου οργανισμού Τελωνίων. με στόχο τα τελωνία να φεγραμμιστούν με τα διεθνή πρότυπα και τι σύγχρονε εμπορικέ πρακτικέ. Αναπτύσσουμε νέα εργαλεία πληροφορική όπως είναι το EU Trader Portal. Ένα άλλο εργαλείο που εξετάζουμε είναι ενιαία θηρίδα για να μπορούν οι οικονομικοί φορείς ηλεκτρονικά και με εναρμονισμένο ολοκληρωμένο τρόπο μία φορά μόνο να εγγράφουν όλες τις πληροφορίες που ζητούνται από την νομοθεσία περί καταναλωτών για τις ε, συναλλαγές ε, της παραδόσης προϊόντων και υπηρεσιών. Θα δούμε και τη μελέτη αντικτύπου, τι αποτέλεσματα θα δώσει για την ε, νέα γενιά προγραμμάτων, για το επόμενο πολιτές μουσομικό πλαίσιο και εδώ έρχομαι στο θέμα που ετέθη για τους ιδίους πόρους, που ήταν και η τελευταία ερώτηση που μου ετέθη. Ο κύριος Μόντι και μια ομάδα εργασία, ο οποίο ηγείτο, κατάρτισε μια έκθεση. Εκπρόσωπος των Γκίφερ Χόφστατ από το Κοινοβούλιο. Δημόσια είναι η έκθεση αυτή και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική εργαλειοθήκη που δείχνει τι έχουμε στη διάθεσή μα για να δράσουμε σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω ότι και οι προτάσεις Μόντι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη, στον πολιτή προβληματισμό χωρίς να αυξηθεί το φορολογικό άχθο. Να έχουμε δηλαδή ίδιους πόρου, πραγματικά ίδιους πόρου, που δεν θα προέρχονται μόνο από τα κράτη. Βέβαια για όλα αυτά θα πρέπει να αναλύσουμε τώρα ποιοι είναι οι πόροι που θα πρέπει να παγιώσουμε και ποιου άλλου θα πρέπει να καθορίσουμε. Δεν μπορώ να σα εκφράσω τι προσωπικέ μου προτιμήσει, αν και θεωρώ ότι ο ΦΠΑ είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Αλλά θα έχω φαντάζομαι την ευκαιρία να σα τα ξαναπώ ή σε εσά και στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Γιατί είναι τόσο αυστηροί οι κανόνες για τους χρήστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι έχουμε το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα από ε, σειρά ετών και αυτό επιτρέπει τελωνιακές απλουστεύσεις και για τον τομέα της ασφάλειας προβλέπονται κάποιες άλλες ε, διατάξεις. Υπάρχει το ΙΕΝΕΣ e και το ΙΕΞΕΣ, e δεν μπορεί να υπάρξει δυνατότητα μη τήρησης των σχετικών ε, προδιαγραφών, όμως βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να πλουστεύσουμε και να διευκολύνουμε τα πράγματα και με συστημικούς ελέγχους. Για τους ε, φορείς AOs, e τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς της Ένωσης τι προστέμενη αξία αναμένουμε από τον κώδικα. Φέρει σημαντικές καινοτομίες, ο εξχωρισμένος θελωνιακός κώδικας και οι όλοι δεσμοί μέτρων που θα επιτρέψει τον εξυγχρονισμό των τελωνιακών διαδικασιών, θα λάβει υπόψη τις σύγχρονες πολιτικές, θα εξορθολογήσει τις διαδικασίες θα επικαιροποιήσει την αρχή του ξεδοτημένου οικονομικού φορέα, θα πλουστεύσει τις τελωνιακέ ε, διατυπώσεις, θα προωθήσει ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί, θα μειώσει το διοικητικό άρθρο για τους οικονομικού φορείς και θα εξασφαλίσει την συνέχεια ε, σε οριζόντιε πολιτικές όπως είναι το ψηφιακό θεματολόγιο και η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τέλος θα εφεγραμμίσει πλήρω το παγκόσμιο περιβάλλον στου τελωνιακού κανόνε, για να έχουμε κοινή δέσμη επικοινωνιακών εργαλείων θα λειτουργούν σε όλη την τελωνιακή Ένωση. Πολύ φιλόδοξο, πολυεπίπεδο αυτό το πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή αγαθών ε, μικρής αξίας, θέλουμε να υπάρξει μαχανοργάνωση των διαδικασιών και διευκόνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Και αυτό έχετε να δέσει με αυτά που είπα πριν για την κυρία Κάλλας που μου είπε οι προτάσεις μας σε ποιο σημείο βρίσκονται για μια οδηγία για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης. Και η κυρία Κάλλας που είναι η συγκίτρια για το θέμα αυτό και έχουμε και την έκθεση της ΙΜΚΟ επί της πρώτης της Επιτροπής για τις κυρώσεις χρηματικές ποινές είναι πολύ σημαντική για την πρόοδο του φακέλου συμφωνώ με τα περισσότερα που λέτε παρά το ότι συνεχίζουμε και τα μελετάμε με προσοχή και όπως ξέρετε η πρόοδος του Συμβουλίου εξαρτάται από το Συμβούλιο και μέχρι τώρα είχαμε πολλές δυσκολίες εκεί γιατί πολλά κρατημένη θεώρησαν ότι ε, μπαίνει στα δικά τους χωράφια το κείμενο αυτό. Και τον Νοέμβριο έγινε συζήτηση στο Συμβούλιο και εννέα κρατημέλη Λοιπόν, θέλω να συνεχιστούν οι συζητήσεις. 12 ήταν κατά για διάφορους λόγους. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει δικαιολογία του να αποσυρθεί η πρόταση. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ζήτηση επί του κειμένου. Άρθρο προς άρθρο. Και περιμένουμε στην ολομελία σας να ψηφίσετε. Οπότε εμεί θα θέλουμε τα κράτη-μέλη να επεξεργαστούν αυτέ τι καθημερινέ γραμμέ με του μου στο εμπόριο. Βεβαίω δεν θα είναι δεσμευτικέ αυτέ τι καθημερινέ. Παρ' όλα αυτά, εάν δεν τι στείλουν τα κράτη-μέλη, τότε εμεί θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία παραβάση. Τώρα για την Τουρκία. Για την Τουρκία είναι θέμα για το οποίο συνεχίζουμε να εργαζόμεθα με τους εκπροσώπους της χώρας της Βρυξέλλας και είμαστε διαθέσιμοι για βελτίωση της τελειωνιακής οικονομικής και οικονομικής συνεργασίας για δε τον Brexit πρόεδρε ε, δεν είναι ότι εγώ επιφυλάσσομαι και διστάζω να το συζητήσω όπως ξέρετε πριν από δύο μέρες άρχισαν διαπραγματεύσει και άρχισαν μόνο μόνο για την δημιουργία πλαισίου, πλαισίου θεματολογίου. Και έχουμε συμφωνήσει όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την προσέγγιση. Άρα δύσκολο να πάμε σε συμπεράσματα. Ακόμα δεν έχουμε συζητήσει τα τελωνιακά. Πάντως υπάρχουν άλλα πολύ δύσκολα θέματα Εγώ πάντως ενδιαφέρομαι και παρακολουθώ από κοντά και προσπαθώ να επερμηθώ των συμφερόντων των αρχών των, των 27 εναντί τη κυβέρνηση της Βρετανίας που θέλει να αποχωρήσει από την Τελωνιακή Ένωση και θέλει άρα να πάει πίσω στον χρόνο πριν την Τελωνιακή Ένωση, τότε που είχαμε τα άκαμπτα, τα σκληρά, τα αυστηρά σύνορα. Δεν είναι δυνατόν. Τι να, να με τέτοιο σύνορο μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Θα πρέπει να βρούμε κάποιες πολιτικές ρυθμίσεις με πρακτικό χαρακτήρα. Ε, αυτή την οτροπία έχουμε ότι θα πρέπει ότι τελικά αν θέλει να βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε κάποιο είδους σχέσεις στενή όσο γίνεται και καλύτερα. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, λέει Πρόεδρο, για τι απαντήσει σα. Δεν ξέρω πώ ακόμα κάποιοι συναδελφοί θέλουν να λάβουν το λόγο. Όχι από ό,τι φαίνεται. Και σας ξανά ευχαριστούμε που ήρθατε. Καλό κουράγιο με τη δουλειά σας. Okay, um, I think we can move... Ωραία, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης που αφορά την παρουσίαση της ε, Κομισιόν ε, σχετικά με τη δέσμη μέτρων ε, για την επιβολή της νομοθεσίας ε, και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην Κομισιόν. το λόγο έχει ο κύριος Ιμφριτ Στρίμαν ο οποίος θα παρουσιάσει το συγκεκριμένο πακέτο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσω το ε, πακέτο εφαρμογής της νομοθεσίας, ε, το οποίο υιοθετήθηκε από την Κομισιόν στις 2 Μαΐου του 2017. Υπάρχουν ε, δύο στοιχεία στο εν λόγω πακέτο, από τη μία το ΣΜΙΤ το άλλο είναι η ε, ε, ψηφιακή ε, πύλη και το άλλο είναι το Solvit. Θα ήθελα λοιπόν να σας τα παρουσιάσω αυτά και θα ξεκινήσω πρώτα με το SMIT, το οποίο είναι το πιο δύσκολο και είναι αυτό το οποίο θα συζητηθεί ιδιαίτερως όταν εξετάζουμε επιχειρήσεις και κράτη-μέλη. Ε, και επίσης επειδή υπάρχουν πολλές παρανοήσεις σχετικά με το τι θέλουμε να καταφέρουμε. Το SMIT είναι ένα εργαλείο το οποίο συλλέγει ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα από τους συμμετέχοντες της αγοράς και γιατί το κάνουμε αυτό είναι επειδή συνειδητοποιούμε ότι ε, επιχειρήσεις θεωρούν ότι η Κομισιόν δεν είναι αρκετά γρήγορη ώστε να ε, περνά τα εμπόδια της ενιαίας αγοράς και πολύ συχνά είναι δύσκολο να συλλεγούν αναλυθούν τα δεδομένα, ούτω ώστε να βρούμε ποιο είναι το πρόβλημα, τη λειτουργία τη αγορά, παραβίαση κανόνων τη ενιαία αγορά ε, και αυτό σε ένα διασυνοριακό πλαίσιο. Πολλέ φορέ τα κράτη-μέλη δεν έχουν επίση τι πληροφορίε ή δεν έχουν την εξουσία να αποκτήσουν τι συγκεκριμένε πληροφορίε, το οποίο είναι μια επιπρόσθετη δυσκολία. Ε, το ΣΜΙΤ λοιπόν προσπαθεί να συλλέξει πληροφορίες όποτε αυτές είναι αναγκαίες ε, για να εξετάσει αν υπάρχει παραβίαση ή δυσλειτουργία στην εσωτερική αγορά. Ε, δεν είναι υποχρέωση έκθεσης, είναι η τελευταία εναλλακτική για την συλλογή πληροφοριών σε ad hoc βάση. Για παράδειγμα, η Ένωση Ευρωπαίων Καταναλωτών παρατήρησε την προστιθέμενη αξία ενός τέτοιου εργαλείου, ώστε η μια αγορά να λειτουργεί καλύτερα για τους πολίτες μας και για τις επιχειρήσεις της ενιαίας αγοράς. Υπάρχουν και ανησυχίες όμως. Το ένα είναι ο διοικητικός άχθος. Ήμασταν προσεκτικοί διότι είμαστε υπεύθυνοι για τις, ε, κυβερ... Ε, για τις επιχειρήσεις ε, και ήμασταν προσεκτικοί ούτως ώστε να μην έχει υπερβολικό διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις. Θα χρησιμοποιηθεί μονάχα σε ορισμένες περιπτώσεις ε, που έχουν ε, σημαντική κοινωνική και οικονομική ε, επιρροή, όπου οι πληροφορίε για την επιχείρηση είναι ο μόνο τρόπο για να συλλεχθούν αυτέ οι πληροφορίε και οι οποίε δεν μπορούν να συλλεχθούν διαφορετικά. Χρειαζόμαστε μια επίσημη απόφαση της Κομισιόν για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο εργαλείο και κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι η Κομισιόν θα συζητήσει πληροφορίε οι οποίε μονάχα είναι διαθέσιμε στην επιχείρηση. Έτσι λοιπόν ω επιχείρηση δεν μπορεί, χρειάζεται να καταφύγει κανεί ε, σε ε, ακριβέ συμβουλευτικέ εταιρείε για να συλλεχθούν τα αναγκαία δεδομένα. Μία άλλη ανησυχία είναι ότι ε, δίνει νέε εξουσίε στην Κομισιόν όλο αυτό. Το SMIT είναι ένα πληροφοριακό εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο ε, των παρόντων μηχανισμών εφαρμογών για τι διαδικασίε επί παραβάση για παράδειγμα δεν θα δημιουργήσει νέες διαδικασίες επιβολής. Ε, παραμένουν τα κράτη-μέλη ε, ε, αυτά τα οποία λαμβάνουν τις πληροφορίες και στα οποία απευθυνόμαστε σε περίπτωση που γίνεται κάποια παραβίαση. Είναι σημαντικό ε, να, ότι, να αναφέρουμε ότι υπάρχει ένα διορθωτικό πρόβλημα σχετικά με τις προφορίες που συλλέγουμε που μπορεί να συνεισφέρουν στη δημιουργία νέων νομοθεσιών εάν είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα ευρύτερο ζήτημα και όχι μόνο ένα στοχευμένο ζήτημα το οποίο αφορά μία και μόνο υπόθεση. Όμω αυτός δεν είναι ο βασικός στόχος. Ο βασικός στόχος είναι να βοηθήσουμε στην εφαρμογή και να χτίσουμε στην, στην, στις υπάρχουσες εξουσίες συλλογής ε, δεδομένων ε, όπου η Κομισιόν εφαρμόζει ε, την νομοθεσία απευθεία στις επιχειρήσεις μέσω των κανονισμών αντιδράσεων. Αυτό, ε, αυτή λοιπόν ήταν η έμπνευση για το συγκεκριμένο εργαλείο και εξετάσαμε το πώς λειτουργούν τα πράγματα σε όλο αυτό. Όμως θέλουμε αυτό να το ε, μεταφράσουμε στους κανονισμούς της ενιαίας αγοράς ούτως ώστε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την ενιαία αγορά ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Έχουμε ε, στην Κομισιόν ε, μια προσέγγιση συνεργασίας με τα κράτη-μέλη που είναι ένα από αυτά τα στοιχεία. Το ΣΜΙΤ το αντιλαμβανόμαστε ως ένα εργαλείο όπου το, η Κομισιόν η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη από κοινού εφαρμόζουν τους κανονισμούς, τα, ε, τους κανονισμούς της ενιαίας χώρας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να ενημερώνονται τα κράτη-μέλη και η πρόταση δημιουργεί μηχανισμούς για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κομισιών και των κρατών μελών Εάν οι πληροφορίε ε, αυτές ακολουθούν μετά από τη διαδικασία επιπαραβάση, τότε η Κομισιόν μπορεί να τα εφαρμόσει αυτά με βάση ε, τις ε, ανησυχίε των κρατών μελών, πέρα από τα δεδομένα όπου οι επιχειρήσεις έχουν χαρακτηρίσει τις πληροφορίες αυτές ως απόρριτες επιχειρηματικές πληροφορίες και τότε δεν είναι υποχρεωμένη να παραδώσει τι συγκεκριμένε πληροφορίε, διότι φοβάται ότι μπορεί να διαρρεύσουν διότι εμεί οι Κομισιόν είμαστε συνηθισμένοι στο να αντιμετωπίζουμε ευαίσθητε πληροφορίε και γνωρίζουμε πώ να τι προστατεύουμε. Και ένα ερώ, τελευταίο ερώτημα στο πλαίσιο του Σμιθ το οποίο εμφανίζεται συχνά είναι για ποιο λόγο ε, έχουμε πρόστιμα, κυρώσει ε, ε, έχουμε παρατηρήσει και με βάση τα μαθήματα τα οποία έχουμε διδαχθεί είναι ότι τα πρόστιμα και οι κυρώσεις είναι ένα κίνητρο ανταπόκρισης. Αυτό είναι το μάθημα το οποίο έχουμε διδαχθεί από την ομοθεσία ανταγωνισμού ε, και ε, σε ε, περίπτωση που ζητήσουμε προφορίες απευθυνόμενοι σε μια αίτηση Smith, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει γίνει κάποιο λάθος αλλά ότι θα πρέπει να υπάρχει μία, αλλά πρέπει να υπάρχει μία απλή αίτηση με εθελοντική συμμετοχή. Ε, υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο εκεί πέρα ε, σε περίπτωση λοιπόν που θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις, ε, τότε θα πρέπει να εκδοθούν τρεις αποφάσεις της Κομισιόν, μία για να ανακοινώσει τη χρήση του ΣΜΙΘ, δεύτερον για να ξεκινήσει η επίσημη αίτηση και τρίτον για την εφαρμογή κυρώσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι για να έχουμε μία απόφαση της Κομισιόν με τόσους πολλούς κομισιό, ε, επιτρόπους ε, θα πρέπει να έχεις καλά επιχειρήματα για να το καταφέρεις αυτό και στο πλαίσιο της νομοθεσίας και των ανταγωνισμού πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν ελάχιστε υποθέσει, οι οποίε όμω θα κάνουν τη διαφορά για την ενιαία αγορά. Είναι ένα εργαλείο τελευταία εναλλακτική, το οποίο θα βοηθ... έρχεται και προστίθεται στην εργαλειοθήκη την οποία ήδη έχουμε για την ενίσχυση τη ενιαία αγορά κατανοούμε ότι ε, όλο αυτό λειτουργεί και είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να εφαρμόσουμε ε, και στον τομέα της ενιαίας αγοράς. Αυτά όσον αφορά το SMIT. Ε, τώρα έχουμε την ενιαία ψηφιακή πύλη, το οποίο είναι το δεύτερο εργαλείο στο πακέτο επιβολής της εφαρμογής της νομοθεσίας. Η πρόταση ε, ήρθε επίσης από εσάς επιχειρήσεις, κοινοβούλιο, μια σειρά κρατών μελών, 17 συγκεκριμένα που ζήτησαν μέσω ε, του ρεφίτ, μέσω ε, των δημόσιων διαβουλεύσεων να υπάρξει κάτι το οποίο θα επιτρέψει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τα ωφέλη της εσωτερικής αγοράς με έναν καλύτερο τρόπο. θα ε, συμβάλλει ότως ε, ε, ώστε να γνωρίζουμε την ομοθεσία των κρατών μελών οι ποιοτικέ πληροφορίε αφορούσαν ε, την βοήθεια ε, που απαιτείται στην εσωτερική αγορά και το ζήτημα έβρεση πληροφοριών, διότι πολύ συχνά υπάρχουν τόσο πολλά δέντρα που στο τέλος χάνεις ε, το δάσος και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται βοήθεια, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τις πληροφορίε που χρειάζονται. επίση το ζήτημα της προσβασιμότητας για Τη προσβασιμότητας σε πληροφορίε για θεσιονεριακούς σκοπού είναι επίση ε, ένα σημαντικό θέμα ε, και επίσης να εξετάσουμε τι εμπόδια υπάρχουν στην εσωτερική αγορά. Ο σκοπό ε, τη ενιαία ψηφιακή πύλη είναι να προσφέρει στου Ευρωπαίου πολίτε και στι επιχειρήσει έναν εύκολο τρόπο χωρί διακρίσει, ούτω ώστε να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίε σχετικά με, την, με του κανονισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών, μελών πώ μπορούν να τηρούν του συγκεκριμένου κανόνε, καθώ επίση και ε, υπηρεσίε βοήθεια για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα δικαιώματά του όσον αφορά την ενιαία αγορά. Η προστιθέμενη, η προστιθέμενη τη ενιαία ψηφιακή ε, πύλη είναι ότι περιλαμβάνει ε, πράξει, δεσμευτικές και μη δεσμευτικές ε, ε, αφορά την ε, πλήρη εφαρμογή. Επιθυμούμε να καλύψουμε τα κενά στην online πληροφόρηση και να συμβάλλουμε σε αυτό για τα κράτη-μέλη αλλά και σε ένα διασυνοριακό πλαίσιο. Επίσης αυξάνει την ποιότητα των ε, πληροφοριών, ε, την ευρυσιμότητα των πληροφοριών, οι όλες οι διαδικασίες αυτές να υπάρχουν online που είναι σημαντικό και να υπάρχει διασυνοριακή προσβασιμότητα. Τεχνικά είναι ε, μια ιστοσελίδα με μηχανή αναζήτησης, με δεδομένα κατανεμημένα σε με βάση κατηγοριοποιημένα ε, έχει έναν μηχανισμό όπου οι χρήστες μπορούν να δίνουν πληροφορίες ε, για να αξιολογείται η ποιότητα. Ε, υπάρχει αυτό το feedback για να μπορέσουμε να βρούμε που υπάρχουν φραγμοί στην ενιαία αγορά. Ε, νομικά τώρα αυτό το οποίο προσπαθούμε να επιτύχουμε με τη συγκεκριμένη πρόταση είναι να αναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να παράσχουν προφορίες σχετικά ε, με διάφορα ζητήματα τα οποία αφορούν ε, πολίτες που μετακινούνται, επιχειρήσεις που θέλουν να λειτουργήσουν διασυνοριακά ε, και συγκεκριμένα πρόκειται για 13 ε, διαδικασίες κλειδιά που θα είναι πλήρως online ε, και θα μπορούν να γίνεται η όλη διαδικασία online για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε ένα άλλο μέλος. Θα υπάρχουν πληροφορίες ούτως ώστε να, γίνεται, να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε όλους τους χρήστες χωρίς διακρίσεις για τις πιο σημαντικές διασυνοριακές διαδικασίες θα πρέπει να υπάρχει η διαδικασία της μίας μόνο φοράς και ότι οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να καταθέτουν τις ίδιες πληροφορίε, ξανά και ξανά, την ίδια γραφειοκρατία, οπότε περιοριζόμαστε σε αυτό. Ε, υπάρχουν κριτήρια για, τις, για τη βοήθεια, για τις αιτήσει ε, και είναι σημαντικό οι προφορίες και οι εξηγήσει ε, για τις διαδικασίες να είναι διαθέσιμες όχι μονάχα στη γλώσσα του κράτους μέλους αλλά και σε μία ακόμα γλώσσα. Αυτή λοιπόν είναι η ενιαία ψηφιακή πύλη, ένα εργαλείο για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουν την ενιαία αγορά με έναν καλύτερο τρόπο. Και το τρίτο από τα στοιχεία ε, του ε, πακέτου είναι το Solvit. Πιστεύω ότι όλοι είστε εκεί με το Solvit. Είχαμε την ικανοποίηση να σας το παρουσιάσουμε στην ΙΜΚΟ πριν από ένα χρόνο, στις 13 Ιουνίου του 2016. Ε, και τώρα, το 2006 και τώρα γιορτάζει τα γενέθλιά του. Ε, είχαμε πάνω από 15.000 υποθέσεις οι οποίες λύθηκαν, ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα, χτίζουμε με βάση αυτήν την ε, επιτυχία και θέλουμε να ε, επεκταθούμε ακόμα περισσότερο συγκεκριμένα θέλουμε περισσότερε επιχειρήσει. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερω από πολίτε, όμω σιγά σιγά χρησιμοποιείται περισσότερο και από επιχειρήσει για ποιο ε, λόγο θέλουμε αυτό το σχέδιο δράσης για να ισχύσουμε το Solvit. Υπάρχει ε, το πολιτικό πλαίσιο. Όταν δημοσιοποιήσαμε τη στρατηγική ε, για την ενιαία αγορά τον Οκτώβριο του 2015 ανακοινώσαμε ότι θα θέλαμε να ενισχύσουμε το Solvit ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη τήρηση των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Και τόσο αυτή η Επιτροπή όσο και γενικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως επίσης και πολλά ενδιαφερόμενα μέλη έχουν ε, εγγραφεί για να ενισχύσουν το Solvit ε, και, με, ε, και κατά συνέπεια η Κομισιόν υιοθέτησε στο πλαίσιο αυτού του πακέτου το σχέδιο δράσης με τρεις πυλώνες που θα βελτιώσει την ποιότητα του Solvit ούτως ώστε να έχουμε καλής ποιότητας πληροφορίες και υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις που απευθύνονται σε αυτό, να αυξήσουμε την χρήση, οπότε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο από ό,τι ως τώρα και στις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να αυξήσουμε, ε, να βελτιώσουμε την εφαρμογή του ε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έχουμε ε, την δήλωση εφαρμογής της Κομισιόν όπου ζητάμε αυτά ο ε, κανόνας να είναι συγκεκριμένος, οπότε θα πρέπει ε, να επικεντρωνόμαστε σε κανονισμούς οι οποίοι είναι οικονομικά πολύ σημαντικοί, οπότε το Solvit βοηθά ούτως ώστε να ε, τηρούνται οι κανονισμοί της ενιαίας αγοράς. Όλες αυτές οι δράσεις πάνε χέρι-χέρι και η επιτυχία του σχέδιου δράσης πράγματι θα εξαρτηθεί από την, ε, από την ορθή εφαρμογή καθενός εξ αυτών ε, και η ε, προϋπόθεση για την, για την επιτυχία είναι να υπάρχει έχει αρκετό προσωπικό το οποίο είναι υποχρέωση των κρατών μελών και ο πιο αδύναμος ε, ε, κρίκος επηρεάζει την συνολική επιτυχία αυτού οπότε το δίκτυο αυτό ε, θα πρέπει να γίνει όσο πιο επιτυχημένο γίνεται ε, θα σταματήσω εδώ λοιπόν και ευελπιστώ στην υποστήριξη αυτής της Επιτροπής ε, σε σχέση με αυτό το σχέδιο δράσης ούτως ώστε να γίνει και αυτό κομμάτι της, ε, του πακέτου επιβολής εφαρμογής της νομοθεσίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σβήμαν για την εξήγησή σας και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους δύο εισηγητές, ένας εξ αυτών είναι η Εύα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ. Συγγνώμη που σα έχω γυρίσει την ε, πλάτη, αλλά ε, τι να κάνουμε εδώ καθόλου. Ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι για την παρουσίασή σα και πρόκειται για προσπάθεια να δώσουμε καινούργια όθηση στην αγορά για υποφελία των επιχειρήσεων αλλά και των καταναλωτών είναι οι βασικές μας μέρημνες. Πασχολούν όλους τους εμπλεκόμενους και ιδιαίτερα τις εταιρείε. Από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι διαπιστώσαμε σε εκείνη την ε, διαβούλευση για το ΣΜΙΤ. Αλλά έχω και κάποιες ερωτήσεις να σας θέσω. Μέσα σε ένα το πρέπει να φύγω, αλλά τέλος πάντων και με συνεργάτε μου πρόκειται να επεξεργαστούμε την απάντησή σα. Οπότε συμπαράτε με, αλλά έχω δυστυχώ μια ταυτόχρονη με την συνάντησή μα υποχρέωση. Οπότε. Για πετε μα, θα ήταν υπερβολικά δαπανηρό οι επιχειρήσει να παίρνουν τις, ε, τις που απαιτούνται από το ΣΜΙΤ και ανησυχώ κυρίως για τις ΜΜΕ Επίσης, πώς εξασφαλίζεται το ότι οι πληροφορίες, τα στοιχεία που δίνουν οι εταιρείε δεν θα στοιχειοθετήσουν ε, υπόθεση εναντίον τους. Ξέρω ότι αυτά τα θεωρείται διαβαθμισμένα ως πληροφορίες, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνουν οι αρχές στα κράτη-μέλη, πώς θα εξασφαλιστεί ότι εκείνες αυτές τις πληροφορίες που θα συλλέξουν δεν θα χρησιμοποιηθούν από ανταγωνιστές ας πούμε ή τέλος πάντων να μην γίνει καμία διαρροή αυτών των δεδομένων. Τέλος, τι μέτρα έχετε λάβει για να καλύψετε αυτές τις ανησυχίες. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις θα υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια να αρθούν οι φραγμοί της ενίας αγοράς. Οπότε Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να είμαστε πιστικοί όσον αφορά αυτή την πρόταση. Να εμπλέξουμε δηλαδή εκείνους. Πέραν του ότι προβλέπονται χρηματικές ποινές για μη υποβολή πλήρων στοιχείων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευαλή Πρόεδρος. Και τώρα, ο άλλος εισηγητής, η άλλη εισηγητρία, μάλλον είναι η κυρία Μίτση που απουσιάζει. Αλλά η κυρία Γιακονσάρη θα μιλήσει στο πόδι της. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν μπόρεσα να είναι εδώ η Μαρλίν δεν κατάφερε να τακτοποιήσει τι υποχρεώσει. της, οπότε τέλος πάντων μου έδωσε εμένα αυτό το σημείο μας το διαβάζω και έχει τις εξή παρατηρήσεις όσον αφορά την πρόταση τη επίτροπή για αυτή την ε, ενιαία ψηφιακή πύλη. Θεωρούμε ότι ακόμα είμαστε σε πρόωρο στάδιο, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο να ε, εξετάσουμε τα πράγματα τα λεπτομέρεια τους. Παρόλα αυτά, καταρχήν αρχήν, θεωρεί την πρόταση της Επιτροπής, ούτως ώστε να θεσπιστεί αυτό το ενιαίο ψηφιακό σημείο εισόδου για υψηλού, υψηλής ποιότητας πληροφορίες για όλα τα διοικητικά και για τις άλλες ε, ε, υπηρεσίες αρρωγής προς πολίτες και επιχειρήσεις. Είναι ψηφιακό ο κόσμος μας και το ίντερνετ και η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζουν τον τρόπο ζωής μας, τον τρόπο που εργαζόμαστε και κάνουμε συναλλαγές, αλλά και ταξιδεύουμε. Είναι απολύτως λογικό, λέει η κυρία Μίτσε, και οι κυβερνήσεις να προσαρμοστούν με αυτόν τον νέο ψηφιακό κόσμο, οπότε να υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες, πληροφορίες και οτιδήποτε ένδικα μέσα, μέσα προσφυγή θέλουν οι πολίτε, οπότε γι' αυτό και είναι κλειδί όσον αφορά το πρόγραμμα δράση η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του κόσμου στον νέο ψηφιακό κόσμο και να δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη για να προσαρμοστούν στις στρατηγικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και έτσι να πάμε σε μια δημόσια υπηρεσία τέτοιου είδους. Πάρα πολύ συχνά ο κόσμος και οι επιχειρήσεις ή δεν, δεν, γνωρίζουν τους κανόνες, σε άλλες χώρες ή δυσκολεύονται να καταλάβουν τις πληροφορίες, τα στοιχεία, τις διαδικασίες που ισχύουν για εργασία, για ταξίδια κλπ. Έχουμε ένα σωρό πύλες, τέτοια σημεία εισόδου, σημεία επαφής για αρρωγή, για τις δεξιότητες και κλπ. Οπότε, αντί να βρίσκουν βοήθεια, τελούν σε σύγχυση οι χρήστες γιατί δεν ξέρουν πού να βρουν την κατάλληλη πληροφορία. Όταν έχουν υπερβολικά πολλές πληροφορίες και σε υπερβολικά πολλά σημεία, αυτό αποτελεί όχι λύση, αλλά φραγμό. Και εμείς πήραμε ένα σωρό αιτήματα για πληροφορία από τον ε, κόσμο. Δύσκολα μπορεί κανείς να βρει σε ένα σημείο όλε τις πληροφορίες που απαιτούνται. Αν υπάρξει ένα τέτοιο σημείο μοναδικό, αυτό θα βγει στον κόσμο. Γι' αυτό και η Μαρλίν θεωρεί ότι είναι θετική προσπάθεια της Επιτροπής που προσπαθεί όλα αυτά να τα μαζέψει. Τις, ε, τα website, τις ε, πύλες, ε, το σημείο εσόδου, ώστε οι επιχειρήσεις, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, ο κόσμος να έχουν φιλικές στο χρήστη πληροφορίες και να βρίσκουν ότι αναζητούν και να αποφασίζουν με τα λόγου γνώσεως. Μηχανισμός που όχι μόνο θα εξοικονομήσει χρόνο, αλλά και χρήμα. Πρώτα θα να σταθεί σε κάποια σημεία η Μαρλίν, αυτά τα οποία θέλει να εξεταστούν ιδιαίτερως. Πρώτα-πρώτα, αυτή η πρόταση θα πρέπει να είναι ένα απλό εργαλείο μέσο για ακριβείς, σαφείς πληροφορίε για πάσα αναγκαία διαδικασία ε, στη χώρα του καθενός ή σε ξένη χώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τίποτα να μην θεωρηθεί ότι αυτό το μέσο αντικαθιστά ισχύουσες διαδικασίες ή νόμους σε εθνικό επίπεδο ή ότι θα μειώσει το επίπεδο προστασίας. Επίσης η Μαρλίνα θα ήθελε να μάθει πώς αποφάσισε η μαρλινα θα ηθελα να μαθει πως αποφασισε η επιτροπη για αυτό τον κατάλογο των 13 σημαντικών διοικητικών διαδικασιών. Έχουμε και άλλες διαδικασίες που προβλέπονται σε κράτη-μέλη. Τι θα γίνει σε εθνικό επίπεδο για αυτές τις άλλες διαδικασίες, πώς θα παρέχονται. Πρότεινε η Επιτροπή να ισχύσει το σύστημα εφάπαξ για την υποβολή των δεδομένων. Να μπορούν να συνεργαστούν αιτήσει του χρήστη και σε διασυνοριακές υποθέσεις. Η Μαρλίν επίσης θα ήθελε να μάθει περισσότερα για τις αρχές που διέπουν το σύστημα. Αν δηλαδή έχουμε υποβολή εγγράφων σε κάποιο κράτος να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ε, έγκυρα τέτοια έγγραφα αλλού χωρίς να υπάρχει διαδικασία ελέγχου του, του, του έγκυρου αυτών και της γνησιότητας. Και να μπορούν επίσης να επικαιροποιούνται έτσι εύκολα αυτά τα έντυπα. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί το ότι πάσα συλλογή δεδομένων θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ασφαλεία να γίνεται σεβαστή αρχή τη προστασία του δυτικού βίου και να υπάρχει αναλογικότητα. Η Μαρίνη προτίθεται να συνεργαστεί αρμονικά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με του πιο δεσηγητέ για την πρόταση αυτή. Ε, ευχαριστώ. Ε, Εμεί ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρο. Θέλει άλλο συνάδελφο τον λόγο για να υποβάλει ερώτηση. Όχι, από ό,τι φαίνεται που θα δώσουμε το λόγο ξανά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με το πρώτο κόστος και δι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη κόστους, αλλά είπα και πριν, είναι ξεκάθαρο για τις ΜΜΕ έχουμε επίγνωση το ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει δυσανάλογο άκθοσες ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας. Άρα τα αιτήματα για πληροφορίες θα πρέπει να είναι πολύ στοχευμένα, ad hoc και θα απευθύνονται μόνο στους συμμετέχοντες στην αγορά που αναμένεται να έχουν στη διάθεσή τους αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή δεν θα στέλνουμε εκατοντάδες επιστολές το αντίθετο. Και θα αφορά η αλληλογραφία δεδομένα που θα είναι διαθέσιμα άμεσα. Απαιτείται δηλαδή περαιτέρω προσπάθεια, παραδείγματο χάρη να προσληφθεί ένα εξωτερικό σύμβουλο ε, για την πρόσβαση στα δεδομένα. Ούτε θα είναι τα ερωτηματολόγια αναλυτικά ε, και διεξοδικά. Θα είναι πολύ συγκεκριμένα τα ερωτήματα. Και ήδη από την αρχή θα περιορίζει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το κόστος των επιχειρήσεων για να απαντήσουν στα αιτήματα αυτά. Και πριν καν ενεργοποιηθεί ένα αίτημα, θα πρέπει να υπάρξει αιτιολόγηση εσωτερικά ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι δηλαδή πράγματι χρειάζεται να υποβληθεί αυτό το αίτημα. Θα το εξετάζω πάρα πολύ προσεκτικά, να δούμε κατά πόσο είναι σκόπιμο ή όχι και αν δεν επιβαρύνει υπερβολικά την επιχείρηση. Επειδή αναφερθήκαμε λοιπόν στις ΜΜΕ, να μιλήσω για τις μικροεπιχειρήσεις που εξαιρούνται βέβαια αυτές. Έτσι. Οι μικρομεσαίες δεν πρέπει να εξαιρούνται γιατί πολύ συχνά τις αφορούν οι δυσλειτουργίες της εσωτερικής αγοράς. Ένα πιθανό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι οι διαδικασίες διαγωνισμών δημόσιων προμηθειών. Μία ΜΜΕ, μια εταιρεία, μπορεί να μην θέλει να δώσει κάποιε πληροφορίε γιατί φοβάται ότι θα την γράψουν σε μαύρο κατάλογο και δεν θα ξαναπάρει ποτέ σύμβαση. Όμως αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν αντιθέτως να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε τα πράγματα που πάνε στραβά και να κινήσουμε διαδικασία επί παραβάση με το κράτος μέλος. Το δεύτερο ερώτημα αφορούσε το απόρριτο, την εμπιστευτικότητα. Πολύ σημαντικό θέμα. Οι πληροφορίες αυτές καθεαυτές δεν δημοσιοποιούνται, είναι σαφές. Το είπα. Υπάρχει το ε, εμπορικό απόρριτο, το επιχειρηματικό, επαγγελματικό απόρριτο, οι επιχειρήσει, μάλλον θα πρέπει αυτές οι υποχρεώσεις να γίνονται σεβαστές και στην προκειμένη περίπτωση. Σε ό,τι αφορά την επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, τις εξουσίες μας τις χρησιμοποιούμε για τη συλλογή πληροφοριών, αλλά μόνο εφόσον αυτό είναι αυστηρά απαραίτητο και με απόλυτη χεμήθεια. και έχουμε ένα μακρό ιστορικό ε, χειρισμού τέτοιων δεδομένων, ευαίσθητων. Αν μια εταιρεία έχει σημειώσει τις πληροφορίες που παρέχει ως ευαίσθητες, αυτό είναι καλό, ε, διότι εμείς θα τις κρατήσουμε τις πληροφορίες και θα τις δώσουμε πουθενά αλλού. Γιατί επιχειρηματικά ε, ευαίσθητες πληροφορίες δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν πουθενά αλλού. Υπάρχει επομένω και ο οικονομικός κίνδυνος γιατί μπορεί κάποιος να πάρει και μήνυση ή να του γίνει καταγγελία, αν δεν τηρεί αυτή την ε, υποχρέωση. Έχουμε εμπειρία από άλλους τομείς και θα τη χρησιμοποιήσουμε και για το εργαλείο αυτό. Διότι αντιλαμβανόμαστε πλήρως δυνητικούς κινδύνους ή θέματα που μπορεί να προκύψουν αλλά το έχουμε στο μυαλό μας. Για την πύλη, την ενιαία. Με χαρά άκουσα ότι η κυρία Μίτσι το υποστηρίζει αυτό το εργαλείο και για την πρότασή μας γενικά τη θεωρεί καλή. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι αυτή η ψηφιακή πόλη ουσιαστικά είναι ένα σημείο στο οποίο φτάνουν όλα τα δεδομένα. Υπάρχουν όμως πολλές διαφορετικές διαδικασίες και τρόποι να πάμε στο επόμενο βήμα. Απλά ξεκινάμε την έρευνά μας από ένα σημείο μόνο. Από εκεί βρίσκουμε όλα τα στοιχεία. Και μπαίνουμε στις δυνατότητες ε, της ενίας από την ίδια πόρτα, αν θέλετε. Γιατί αυτό που λείπει είναι πολλές φορές ότι ενώ ξέρουμε ότι υπάρχουν τα στοιχεία, δεν ξέρουμε πού να τα βρούμε. Θα διευκολύνει αυτό και τις διασυνοριακές διαδικασίες, καθιστώντας τις λειτουργικές. Και αυτό είναι προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Θα είναι ως το δυνατόν πιο απλό το σύστημα, αυτή είναι η πρόθεσή μας και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των προσπαθειών μας σε όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή θέλουμε να προωθήσουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλα τα κράτη-μέλη. Και με αυτή την ενιαία ψηφιακή πύλη θα βοηθήσουμε σε κάποια κράτη-μέλη, όχι μόνο για τα δύο συνοριακά, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, εθνικό επίπεδο, γιατί πολλές χώρες μέλη δεν είναι προχωρημένες σε αυτές τις διαδικασίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Άρα όλοι κερδισμένοι θα βγουν και οι εγχώρες επιχειρήσεις. που θέλουν να δραστηριοποιηθούν και εκτός των εθνικών σύνορων και διασυνοριακά. Θα μπορέσουμε να ξυγχρονίσουμε την ε, λειτουργία των ε, διοικήσεων. Φυσικά και θα ήταν ανόητο τα έγγραφα ή τα στοιχεία να χρειάζεται κανείς να τα εισαγάγει παραπάνω από μία φορά. Γι' αυτό θέλουμε αυτό να γίνεται μία φορά μόνο. Σίγουρα μπορεί να προκύψουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Πάντοτε υπάρχουν δυσκολίες. Ιδίως αν υπάρχουν ε, σε ισχύ διαδικασίες και αν κάποιοι δεν θέλουν να τις ε, εγκαταλείψουν. Γιατί παρότι και αν, παρότι και αν μπορεί να είναι καλύτερο το νέο σύστημα υπάρχει μια αντίσταση συνήθως. Πρέπει λοιπόν να πείσουμε και τους λιγότερο ενθουσιώδεις να ακολουθήσουν Θέλουμε να υπηρετούμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ουσιαστικά και όχι τις επιχειρήσεις, ε, και όχι να δημιουργούμε προβλήματα. Εδώ ολοκληρώνω, βέβαια είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σβήμαν. Δεν νομίζω ότι θέλει κάποιος να σας κάνει συμπληρωματική ερώτηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά που ήρθατε στην Επιτροπή μας και μας εξηγήσατε το πακέτο συμμόρφωσης. Με αυτά και με αυτά μπορούμε να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, εφόσον είναι εδώ η ό,τι μου λένε, μάλλον θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο. Να έρθει εδώ ο εισηγητής, κύριος Βάντεν Χόλτσερ, ή κάποιος άλλος τέλος πάντων. Ας κάνουμε δύο τρελατά διάλειμμα. Πέντε παρατέταρτο ξανά θα ξεκινήσουμε. Okay, uh, I think we can... Uh, Ωραία, πιστεύω ότι ε, μπορούμε να αρχίσουμε ή να συνεχίσουμε μάλλον ε, με το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης για σήμερα ε, που αφορά την το σχέδιο δράσης για τις ε, λιανικές ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ε, και καθώς ο κύριος Βάιντεν Χόλτσα δεν είναι εδώ θα μιλήσει εκ μέρους του. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δυστυχώς δεν είναι ανάμεσα μας ο Γιώζαφ και μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω, κάτι το οποίο κάνουμε μεγάλη ευχαρίστηση. Ε, και ε, πολύ απλά θα διαβάσω το κείμενο το οποίο ε, μου έδωσε, το οποίο αφορά την γνωμοδότηση για ένα σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πρότασή της για το σχέδιο δράσης για τις ελληνικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ε, το σχέδιο δράση που παρουσίασε η Κομισιόν αντικατοπτρίζει τα ε, σχέδια τα οποία ε, το Κοινοβούλιο παρουσίασε στην Πράσινη Βίβλο του και όπου συμμετείχε και η ΙΜΚΟ. Παραδείγματα για αυτό είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις, ε, στα τέλη για τις διασυνοριακές συναλλαγές, την ηλεκτρονική υπογραφή, ε, Παρ' όλα αυτά όμως το σχεδικό δράσης ε, παραμένει ε, γενικό λογό και ε, απαιτείται μια πιο καλή παρακολούθηση της αγοράς και εμείς ως Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ζητήσω στις επιχειρήσεις που είναι διασυνοριακές να, υπά... να αναφέρεται τόσο η τράπεζα της χώρας προέλευσης όσο και υποδοχής. Επίσης θα πρέπει ε, να αναφέρεται ε, και ε, το ζήτημα των των συναλλαγμάτων ε, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι πάνω σε αυτό. Η ηλεκτρονική υπογραφή ε, θα μπορέσει να βοηθήσει σε πιο ασφαλείς διασυνοριακές πληρωμές ε, εφόσον όμως το ίδιο το σύστημα είναι ασφαλές και η ηλεκτρονική ταυτότητα και κλοπής αυτής είναι κάτι το οποίο αποκλείεται. Επίσης η ηλεκτρονική υπογραφή δεν θα πρέπει να οδηγήσει ούτως ώστε οι χρήστες να μην μπορούν ή να μην θέλουν να χρησιμοποιήσουν υφίσουν αυτό το πρόγραμμα ή να ε, ε, υφίστανται διακρίσεις. Ε, η γνωμοδότηση είναι αρκετά σύντομη και μέχρι τις 29 Ιουνίου θα υπάρξουν τροπολογίες και θα γίνει πιο συγκεκριμένη και μετά το διάλειμμα του καλοκαιριού θα ακολουθήσει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Προσβλέπω στη συνεργασία με τους σκιώδεις και εμείς ε, ε, ευελπιστώ να περιλάβουμε την ε, έκθεσή μας στην έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Εύελιν, που μίλησε εκ μέρους του κυρίου Βάιντενχόλτσα. Υπάρχει κάποιος άλλος, ίσως ο κύριος Πόσφιζιλ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ θα μιλήσω εκ μέρους ε, του EPP. Ε, ε, εξετάσαμε λεπτομερώς κείμενο το οποίο κατέθεσε ο κ. Βάιντεν Χόλτσερ και χαιρετίζουμε τη συζήτηση για ε, την νομοθεσία που ε, καθιστούν ε, πιο εύκολες τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για τους πελάτες, όμως αρχικά θα θέλαμε να εξετάσουμε την νομοθεσία στα μεμονωμένα κράτη-μέλη και να εξετάσουμε αν το εθνικό δίκαιο είναι προβληματικό και σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβαίνει τότε ε, θα πρέπει ε, να εξετάσουμε τα ε, δευτερεύοντα δικαιώματα τα οποία αφορούν το ζήτημα αυτό. Αν υπάρχουν τέτοια προβλήματα τότε θα μπορούσαμε ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κινηθούμε. Είμαστε κατά ε, του ε, να υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια νέα νομοθεσία και να, που θα επεμβαίνει στο εθνικό δίκαιο. Σε εθνικό επίπεδο λοιπόν αρχικά θα πρέπει να γίνει η ανάλυση εάν ε, υπάρχουν κάποια προβλήματα ε, και ε, στην συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσουμε το την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης ε, τα ζητήματα τα οποία αφορούν την φορολογία αλλά και τη γλώσσα θα πρέπει να τα σεβαστούμε, δεν θέλουμε αυτά να ε, καταργηθούν μέσω μιας νέας ε, νομοθεσίας ή οδηγίας και γι' αυτό το λόγο τα βλέπουμε όλα αισιόδοξα όμως αρχικά θα πρέπει να ρυθμιστεί αν υπάρχει ανάγκη για μια νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ε, θέλουμε ε, λοιπόν η ε, αρχή της αναλογικότητας και της επικουρικότητας να τηρηθεί. Επίσης θα ήθελα να μιλήσω για το κείμενο. Δυστυχώς όμως ο εισηγητής δεν είναι εδώ, οπότε δεν έχει νόημα να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για μια συνάντηση με τον κύριο Βάιντενχολτσα ε, όμως υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε. Ε, αρχικά ε, δεν θέλουμε να υπάρχουν σημαντικά τεχνικά προβλήματα με το, κύμα, ναι, με το κείμενο. Θα πρέπει να υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία αφορούν την γλώσσα. Επίσης την τα, όσον αφορά τα εμβάσματα Αυτά θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Επίσης, ποιοι είναι οι παράγοντες που συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ε, σε αυτό το θέμα θα θέλαμε ε, μία ε, μία πιο συγκεκριμένη πληροφόρηση από τα κράτη-μέλη. Επίσης υπάρχει ο λόγος ε, για μια ε, πιστοποίηση. Στο παρελθόν επανειλημμένα ήμασταν κατά της εισαγωγής πιστοποιητικών και θα θέλαμε να μάθουμε πώς το εννοεί ο γνωμοδότης αυτό υπό το άρθρο 5 ε, και για το αν θα πρέπει να εισηχθεί μια υποχρεωτική ε, ε, πιστοποίηση. Στο σημείο 6 αναφερόμαστε στην ε, ηλεκτρονική υπογραφή η οποία θα πρέπει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να, να λαμβάνουμε υπόψη και για τον κίνδυνο κλοπής της ηλεκτρονικής ταυτότητας και Γι' αυτόν τον λόγο, ε, όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα θέλουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Βάιντεν Χόλτσα, οπότε πιστεύω ότι μπορούμε να εργαστούμε πάνω σε αυτό, προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πόσπισιλ. Υπήρχε μια καθυστέρηση με τη μετάφραση. Είδα ότι και εσείς θα θέλατε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρους της Άλντε θα ήθελα να ε, κάνω κάποια ε, σχόλια. Όμως, καταρχάς, καλώς ήρθατε στην πρώτη σας ε, μέρα. Ευελπιστώ ότι όλες σας οι ως Πρόεδρες θα είναι τόσο σύντομες όσο η σημερινή. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την γνωμοδότησή του. Πιστεύω ε, είναι κρίμα που δεν είναι ανάμεσά μας. Ε, όπως και να έχει, οι συνάδελφοί μου αναρωτιούνται αν υπάρχουν προβλήματα ε, σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές ε, υπηρεσίες. Ε, σας διαβεβαιώνω ότι εμείς βλέπουμε αρκετά ε, προβλήματα. Η πλειονότητα των ε, Ευρωπαίων πολιτών, 92% δεν έχουν αγοράσει κανένα από, καμία από αυτές τις υπηρεσίες στη χώρα τους, οπότε ναι το βλέπουμε ως πρόβλημα. λιγότερο από ένας στους 20 ε, των ερωτηθέντων αγόρασαν, ε, έκαναν τον ε, τραπεζικό τους λογαριασμό, την πιστοτική τους κάρτα σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο κατοικούν, οπότε βλέπουμε, θεωρούμε ότι πρόκειται για μια ανεξερεύνητη αγορά που δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά και σίγουρα το θεωρούμε ένα ε, πρόβλημα και παρόλο που βλέπουμε την στάση αν έχει ένα τραπεζικό λογαριασμό σε άλλη χώρα και το πεις σε κάποιον τότε σε αντιμετωπίζουν λίγο πολύ σαν να είσαι εγκληματίας. Έχω, λογαριασμό σε άλλη χώρα και θα σου πούν ότι περίεργο. Είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτή... Έχουμε αυτή την αντιμετώπιση. Ε, που δεν υποστηρίζουμε καθόλου την ομοθεσία την οποία προσπαθούμε να ε, εισάγουμε. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να γίνει κάτι πάνω σε αυτό. Χαιρετίζουμε το σχέδιο δράσης το οποίο έχει προταθεί από την Κομισιόν, όμως ε, βλέπουμε κάποια θέματα τα οποία θα θέλουμε να τονίσουμε πρώτον τις, ε, τους περιφερειακούς αποκλεισμούς ε, που το συζητήσαμε σε άλλες επιτροπές, το υποστηρίζουμε ιδιαιτέρως ε, ότι θα πρέπει να καταργηθούν. Ευελπιστούμε να υπάρξουν σύντομα λύσεις στις διαθεσμικές συζητήσεις και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει μια λύση πάνω σε αυτό. Ε, επίσης όσον αφορά τις δυσυνοριακές ε, συναλλαγές, ε, αυτό είναι ένα μυστήριο. Δουλεύω εδώ στο Κοινοβούλιο και έχουμε χρήματα από ένα σουηδικό λογαριασμό προς το Βέλγιο και από το Βέλγιο προς, το, προς τη Σουηδία και ποτέ δεν ξέρω πόσο είναι τα τέλη για αυτό. Το κάνω διότι μπορώ να το κάνω, όμως φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι το να στέλνουμε ε, χρήματα χωρίς καθόλου τέλη. Μερικές φορές ε, με ρωτάνε ε, θέλετε να το κάνετε και αποδέχεστε τα τέλη. Εγώ κλικάρω ναι. Δεν ξέρω όμως πόσο είναι αυτά τα τέλη, το οποίο είναι απίστευτο. και θέλουμε πρώτα να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο και στη συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, ίσως ε, επειδή έχουμε ε, δει τις αλλαγές θα θέλαμε να λάβουμε υπόψη την οδηγία πληρωμών και θα θέλαμε να προχωρήσουμε πάνω σε αυτό και τέλος όσον αφορά την ψηφιακή κοινοτομία για τις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες βλέπουμε τα παραδείγματα τα οποία θέλει να εισάγει η Κομισιόν και για τη χρήση ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που ε, παραμένει περιορισμένη σε εθνικό επίπεδο και γι' αυτό το λόγο υποστηρίζω αυτή τη βούληση και θα ήθελα η Κομισιόν να το ε, προωθήσει. Ε, το επόμενο βήμα λοιπόν θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα ούτως ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση όταν προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία. Αν Ανυπομονώ λοιπόν να ε, συνεχιστεί ο διάλογος και σίγουρα θα καταθέσουμε τρομολογίες με βάση αυτά τα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ε, δεν βλέπω κάποιον άλλον. Ε, δεν ξέρω, Εύελιν, αν εσύ θα ήθελες να απαντήσεις. Συγγνώμη, πρώτα η Επιτροπή. Ο κύριος Τσέικοπ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομο θα είμαι γιατί βλέπω ότι υπάρχει κάποια υποστήριξη αυτό το σχέδιο δράση Εν συντομία, σε σχέση με ορισμένε από τις δράσεις, ε, θα ήθελα να πω ότι Έχουμε ξεκινήσει το διερευνητικό μας έργο και θα δρομολογήσουμε διαβουλεύσεις, για παράδειγμα, σε σχέση με το πώς μπορούμε να μειώσουμε το κόστο των διασυνοριακών συναλλαγών και η μετατροπή των νομισμάτων ε, να είναι πιο διαφανής ε, σε ό,τι αφορά το ε, θέμα της ισοτιμίας αναφοράς, του επιτοκίου αναφοράς. Και σε ό,τι αφορά τα εμπόδια στη διασυνορική παροχή υπηρεσιών, Και εδώ ακολουθούμε μια διερευνητική προσέγγιση γιατί γνωρίζουμε ότι είναι μικρής σε οι διασυνοριακές υπηρεσίες που παρέχονται. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στις πολύ διαφορετικές νοοτροπίες ε, και κουλτούρες σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών μεταξύ άλλων. Συνεργαζόμαστε με τους ενδιαφερομένους φορείς και τα κράτη-μέλη για να δούμε πού έγκυνται τα εμπόδια Ξεκαθαρίζουμε επίσης ότι θέλουμε να παραμείνουν υψηλά τα επίπεδα προστασίας των καταναλωτών, άρα σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να υποβαθμίσουμε τα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών. Κάποια άλλα ζητήματα που αναφέρατε περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης, εδώ όπως είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα. Και φυσικά οποιαδήποτε υποστήριξη των δράσεων που έχουμε αναγγείλει είναι καλοδεχούμενη αν θέλετε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, με τα χαρά να το σημειώσουμε και να δούμε βέβαια στην πράξη τι μπορούμε να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά το χρονικό ορίζοντα για αυτό το σχέδιο δράση. είναι μια διετία, αν προσέξατε τις δράσει που επισυνάπτονται στο κατάλογο. Σίγουρα δεν πρόκειται όλα αυτά να λύσουν ε, οριστικά ε, το ζήτημα και να έχουμε μια ολοκληρωμένη αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αλλά κάνουμε ένα βήμα. Ευχαριστώ πολύ προ τον κύριο Τζέικοπ και ίσως κάποιες καταληκτικές πατήσεις από την κυρία Γκέπχαρτ. Ναι, ευχαριστώ. Ε, πράγματι είναι κρίμα που δεν είναι ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ εδώ για να δει και πόσο σοβαρά λαμβάνεται υπόψη η δουλειά. Τέλος πάντων, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό για τη δική μας Επιτροπή εδώ, τομέας της προστασίας των καταναλωτών, Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, ξέρουμε ότι ασχολείται με τα λεπτομεριακά ζητήματα που αφορούν τις χρηματικές συναλλαγές, όλα τα οικονομικά θέματα, τα γνωρίζει άλλωστε. Πάντοτε όμως η εμπειρία μας μας δείχνει ότι η πτυχή προστασίας του καταναλωτού ε, πέφτει σε δεύτερο πλάνο και γι' αυτό εμείς ως Επιτροπή έχουμε το καθήκον να θέτουμε αυτά τα ζητήματα και σε ό,τι αφορά τον πρόσωπο της ΑΛΔΕ Πραγματικά είπατε πολύ σωστά ότι πολύ συχνά ε, όταν γίνονται οι συναλλαγές δεν ξέρουμε ποια είναι η ισοτιμία ε, μετατροπής και όταν δεν είναι το ευρώ δηλαδή, το νόμισμα. αν κάποιο θέλει να κάνει ε, διακοπές, ε, δεν έχει πολλά λεφτά και θέλει να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, ε, θέλει να το πληρώσει των προτέρων γιατί αυτό είναι πιο φτηνό, δεν ξέρει πόσο θα κοστίσει και ποια τράπεζα τελικά απαιτεί τα τέλη της διασυνοριακής συναλλαγής. Δεν μπορεί κανείς να επιλέξει δηλαδή με γνώσεως. Δεν διευκολύνει το καταναλωτής. Τέτοια θέματα ε, πρέπει νομίζω να μας απασχολήσουν. Οι ερωτήσεις τώρα πετέθησαν ε, επειδή δεν είναι για μένα αλλά για τον ε, συνάδελφο. Δεν μπορώ εγώ να ερμηνεύσω. Έχει το συνεργάτη του εδώ ο συνάδελφος που έχει σημειώσει τα ερωτήματα και φαντάζομαι ότι είτε διμερός είτε σε μια συνάντηση μεταξύ του εισηγητή και των σκιωδών θα μπορέσουν να λυθούν όλες οι απορίες. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Evelyn. Ευχαριστούμε πολύ, Evelyn. Νομίζω ότι αυτέ ήταν οι τελευταίε παρατηρήσει για αυτό το θέμα τη μέση διάταξη. Μπορούμε επομένω να το κλείσουμε. Α, και ευχαριστώ που μου το υπενθυμίζετε. Η προορισμοί για τι τροπολογίε είναι η 29η Ιουνίου. Όλοι παρακαλώ να υποβάλουν τις τροπολογίες τους μέχρι τότε. Οπότε θα γυρίσω το πέρας αυτής της ε, συνεδρίασης. Ευχαριστούμε τους διερμηνές Και ευχαριστούμε και την γραμματεία. Θα αρχίσει σε περίπου μισή ώρα η συνεδρία των συντονιστών.